η ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Η επόμενη συνεδρίαση αύριο, 5η 18 Απριλίου, από τις 9 ε, μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 5. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και έχει αναρτηθεί στο ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού